Je vous remercie de prendre place. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να α, πάτε στις θέσεις σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και εσείς οι διερμηνείς. Θα περάσουμε αμέσως στην ημερήσια διάταξη που α, σας μοιράστηκε. Σας ζητώ λοιπόν να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Επίσης έχετε, έχετε τα πρακτικά της συνεδρίασης online, της προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, θα ήθελα να εγκριθούν τα πρακτικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στα πλαίσια της εβδομάδας περιφερειών η Επιτροπή μας αλλά και η Επιτροπή θα οργανώσουν την, την ετήσια συνεδρίαση, η οποία θα ε, προεδρεύεται από την κυρία Ιζαμπέλ Μποντινό, που συνάντησα ε, αμέσως μετά την εκλογή μου, και τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ρεγκή. 3 Οκτωβρίου από τις 9 η ώρα στο χώρο της Επιτροπής Περιφερειών Προφανώς ε, είστε ευπρόσδεκτοι και ε, σας προσκαλούμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ο Επίτροπος ε, Ζώνας Αλ, που είναι ακόμα υπεύθυνος της πολιτικής συνοχής μέχρι τον Οκτώβριο, θα συμμετάσχει στη συζήτηση μαζί μας και θα συζητήσει την εφαρμογή των κονδυλίων. Σας προσκαλώ λοιπόν για αυτή την συζήτηση και ελπίζω ότι οι εργασίες μεταξύ των δύο ε, επιτροπών θα αποδώσουν καρπούς. Όπως πάντοτε ήταν καρποφόρες μάλιστα. Θα ήθελα να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσης διάταξης όσον αφορά στην ψηφοφορία του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό του 2020. Θα ήθελα λοιπόν να πάρετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας, να τις ε, ε, περάσετε στη μηχανή. 40 μία τροποποίησης συζητήθηκαν μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Είσαστε έτοιμοι για να ψηφίσετε. Μιλάω για, αναφέρομαι στα καινούργια μέλη που ενδεχομένως μπορεί να έχουν κάποιες απορίες. Συμβιβασμός 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχή ή εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροποποίηση 10. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. 13. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Τροποποίηση 3. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. 14. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. 15. Υπέρ, κατά, Εγκρίθηκε. Συμβασμό 3. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Αποχή, κανένας, άρα εγκρίθηκε. τροποποίηση του εισηγητή, προφορική τροποποίηση του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Τροποποίηση 18, υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Τροποποίηση 19. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Συμβασμό 4. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Συμβασμό 5. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Όσον αφορά στην τροποποίηση 24, με την προφορική τροποποίηση που κατατέθηκε από το ΕΛΚ υπέρ κατά αποχή εγκρίθηκε. Τροποποιητική 10 υπέρ για τον συμβιβασμό 6. Υπέρ κατά αποχή εγκρίθηκε. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχή εγκρίθηκε. Στο 8 υπέρ κατά αποχή εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροποποίηση 33. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Στο δεύτερο κομμάτι της ε, τροποποιητικής 33, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε σε επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 ε, υπέρ, 16 κατά. Το δεύτερο κομμάτι εγκρίθηκε. Τροποποιητική 36 υπέρ, κατά, αποχή, απορρίφθηκε. Τροποποίηση 39. Κατά, υπέρ, κατά, αποχή, απορρίπτεται. Τροποποιητική 40 υπέρ αποχή κατά Τροπολογία 40 Άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 22 κατά, υπέρ 8, απορρίπτεται. Τροπολογία 41, υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίθηκε. Παίρναμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Σχεδόν ομόφωνα. Σε Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Περνάμε στο σημείο 5. για την συνέχιση των ε, ε, διαπραγματεύσεων για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπω γνωρίζετε ξεκίνησαν ε, την προηγούμενη θητεία οι συζητήσεις με τρει τριμερεί, ε, το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Κατά την ε, τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας επιβεβαιώσαμε την συμμετοχή τη συμμετοχή των συναδέλφων ως, ως συνεισηγητές του κ. Νοβάκοφ και Κρέλ. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Θα συνεχιστούν ε, πολύ γρήγορα, ε, αν δώσετε και την έγκρισή σας, αύριο το απόγευμα. Το άρθρο 52 του κανονισμού προτείνει την ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου θα είναι η αρχή στη βάση της συνεργασίας. Κατά, πλειοψηφία τα μέλη μπορούν ε, να ε, συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε στις, ε, στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, γνωρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν δεν έχουμε κατελάχιστο ε, υπέρ την ψήφο 22 ε, βουλευτών της ε, Επιτροπής. Θα ζητήσω λοιπόν από τον εισηγητή να πάρει το λόγο πριν συνεχίσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Νοβάκοφ έχει το λόγο και η κυρία Σονσουέζ μετά να έχει το λόγο. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την άρεξη των αντιπραγματεύσεων. Αυτό που πετύχαμε στη Ρουμανική Προεδρία να το συνεχίσουμε. Υπάρχει και η χρονική πίεση να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε άμεσα. Να μας δώσετε λοιπόν την εντολή. Σε λιγότερο από 12 ώρες μπορούμε να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με την Προεδρία και την Επιτροπή. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που Τα μπλοκ 1, 2 και 5 είναι πολύ σημαντικά για τη, για τη Φιλανδική Προεδρία, ώστε να οι περιφέρειες να ξεκινήσουν με, το, με τον προγραμματισμό. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ τόσο με την θέση του συνεισηγητή. Είχαμε άτυπες συζητήσει ε, θετικές και οι οποίες μας επιτρέπουν, νομίζω, να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις πολύ σύντομα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην ε, ηλεκτρονική ψήφο επί του εξής. Είστε υπέρ της επανάληψης των διαπραγματεύσεων για τις κοινέ διατάξεις, δηλαδή του CPR. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ, ψηφίστε. Le vote Πέρας. 37 υπέρ, 4 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές, με συγχωρείτε, και καλή επιτυχία στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Ο επόμενος τριμερής διάλογος είναι για αύριο, το είπα ήδη. Να είστε σίγουροι ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης ε, θα υπερασπιστεί αποφασιστικά την ε, πολιτική συνοχή για τα 7 επόμενα έτη. Ακριβώς έτσι θα προχωρήσουμε και για το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 52 άρθρο του κανονισμού, προλέπει τα εξής ότι η θέση που θα έχει υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστά την εντολή για όλες τις διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Και ότι η αρμόδια επιτροπή μπορεί να βασίσει διαπλειοψηφίες να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ακολούθως. Οι συνεισηγητές ο Ανδρέα Κοτσολίνο θα ήθελε το λόγο προτού προχωρήσουμε στην ψήφο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι είναι σημαντική η ψήφος για τις ερχόμενες εβδομάδες ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε τις εξακριβώσεις που χρειάζονται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε στην ψήφο. Παρακαλώ, ψηφίστε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Επομένω, το συντομότερο δυνατό μπορούμε να επανέλθουμε στι διαπραγματεύσει. Συγχαρητήρια στου συνεισηγητέ και επίση και εδώ προφανώ καλή επιτυχία για τη διαπραγματεύση στο ΦΕΝΤΕΡ. Πολύ σημαντική και συνδεδεμένη με εκείνη του CPR. Λοιπόν, αν συμφωνείτε δεν θα επανέρχομαι κάθε φορά στην πλήρη περιγραφή της διαδικασίας. Με τον ίδιο τρόπο προχωρούμε για τον κανονισμό της εδαφικής συνεργασίας Interreg. Πασκάλ αριμό παρακαλώ, έχετε το λόγο αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, αλλιώς θα περάσουμε απευθείας στην ψήφο. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Να παρακαλήσω τους συνδελφούς να συμφωνήσουν συμφωνήσουν για να προχωρήσουμε στην τριμερή διάλογο στο δυνατόν πιο γρήγορα. Bien. Donc nous allons procéder. Καλώς. Ψήφος. Αποδέχεστε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τον κανονισμό Interreg. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Ομοφόνος. Να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στους ρημότερο δυνατών. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον εισηγητή. Το ίδιο για το μηχανισμό άρσης των εμποδίων, λέει ο πρόεδρος των νομικών και των διοικητικών σε διασυνοριακό πεδίο. Χριστιαν Κινέα, ο ηγητής, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια για να πάμε στην ψήφο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά να συνεχίσω την προηγούμενη δουλειά στον φάκελο αυτό που είναι σημαντικός. Ε, προσπαθώ να διευκολύνουμε την ζωή των ε, πολιτών και των επιχειρήσεων όπως και των αρχών στις διασυνοριακές περιφέρειες. Ε, θα σας διατηρώ ενήμερους εγώ και η ομάδα για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ, λέω Πρόεδρος. Πάμε να ψηφίσουμε λοιπόν στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο επί του κανονισμού αυτού. Παρακαλώ, ψηφίστε. Le vote est clos. Πέρασε. Έχετε την εξουδότηση λοιπόν από την Επιτροπή. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Αντιστοίχω, για την επανεκκίνηση των επαναπατεύσεων, για την προχρηματοδότηση, την ετήσια, για τα έτη 2021 έως 2023, η κυρία Μοσαντόφσκα αν θα επιθυμούσε να μας πει δύο λόγια πρωτού προχωρήσουμε τη ψήφο. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ την ε, υποστήριξή σας για την εντολή διαπραγμάτευσης. Ε, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να περάσει στους ε, τριμείς διαλόγους. Δεν έχουμε ακόμα τη θέση συμβολίου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και θα πρέπει ε, στα ακόλουθα τρία χρόνια να έχουμε τις απαραίτητες ποσοστώσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ουσιαστικό τη σημασία σημείο. Ε, θα ήθελα την υποστήριξή σας για την εντολή διαπραγμάτευσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέω, ο για τις εξηγήσει αυτές. Πάμε λοιπόν στην ψήφο για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων, παρακαλώ ψηφίστε. Le vote est clos. Πέρας. Υπάρχει λοιπόν εξοδότηση διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον εισηγητή. Σημείο 10 τώρα. Τι ημισής διατάξεως για την χρηματική στήριξη προς τα κράτη-μέλη λόγω του διοικητικού άχθους, λόγω της πιθανής έτσι, αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ατάκτους που λέμε. Επί της αρχής και λέγω επί της αρχής 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει όπως αντιλαμβάνεστε κανενός είδους βεβαιότητα δεδομένου, δεδομένου του πολιτικού πλαισίου, του πολύ ρευστού. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προβλέψει κανείς τι ακριβώς θα συμβεί στο τέλος του μήνα. Θα έχουμε συμφωνία ή μήπως θα έχουμε no deal. Κανείς δεν τολμά να τοποθετηθεί με εκτιμήσεις. Εμείς όμως οφείλουμε να προετοιμαστούμε για μια άτακτη αποχώρηση, no deal, που θα ενείχε πολύ σημαντικές δυσκολίες και περιπλοκές, όπως και χρηματικές επιπτώσεις για διάφορες περιφέρειες και κράτη-μέλη που έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς οικονομικούς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ώστε να έχουμε ένα μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να ενισχύουμε, να βοηθούμε τις περιφέρειες, τις περιοχές εκείνες των κρατών μελών που θα είχαν τον υψηλότερο αντίκτυπο. Επομένω υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Μία που σχετίζεται με την άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και που θα προέβλεπε το υποθετικό σενάριο του να μην έχει πλέον πόρους στο Ταμείο γιατί αυτή τη στιγμή καλείται να καλύψει τις φυσικές καταστροφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένω προβλέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να ζητήσουν από αυτό το νέο σκέλος του Ταμείου για τα έτη 2019 και 20 μόνον, μόνον από 1η Νοεμβρίου 2019 αντισταθμίσεις, αποζημιώσεις, οι οποίες θα ήταν δυνατές μόνον μέχρι το τέλος του 2020 και μόνον μέχρι το 50% του προϋπολογισμού του συνολικού του Ταμείου. Τα υπόλοιπα προφανώς εξακολουθούν να είναι αποθεματικά έναντι φυσικών καταστροφών. Η δεύτερη υπόθεση που σχετίζεται, η δεύτερη διάσταση που σχετίζεται με το Brexit είναι η αύξηση από το 10% στο 25% των κονδυλίων του Ταμείου, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις προκαταβολές, λοιπόν, οι οποίες θεωρούνται αυτή τη στιγμή μη επαρκείς και οδηγούν σε καθυστερήσει στο έδαφο μετά από επιπτώσει φυσικών καταστροφών. Η Επιτροπή Προπολογισμού εξέτασε την πρόταση αυτή και μας διαβίβασε μια γνωμοδότηση η οποία είναι θετική. Την έχετε λάβει. ...5 Σεπτεμβρίου ο κίνδυνος της άτακτης αποχώρησης ήταν εξαιρετικά υψηλός 5 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, εξακολουθούμε να πλέουμε σε απολύτως άγνωστα ύδατα. Μεταξύ της 5 Σεπτεμβρίου και της σημερινή ημέρας, κάπως κινήθηκε το πράγμα και καθόλου δεν γνωρίζουμε ότι πράγματι θα υπάρξει η αποχώρηση την 31η Οκτωβρίου. Είναι λοιπόν, όπως έλεγα, άγνωστα τα ύδατα και η κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναβάλει την εξέταση του χαρτοφυλακίου αυτού μέχρι ότου το πλαίσιο του Brexit αποσαφινιστεί. εφόσον έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις, μπορεί το πράγμα ξαφνικά να καταστεί υπερεπίγον. Κάποια κρατημέλη στο Συμβούλιο επιθυμούν να τροποποιήσουν ως προς τα όρια την πρόταση, όρια δηλαδή ανά των οποίων θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει δυνατότητα να κινηθεί ταχύτατα αντιθέτως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο υπόκειται σε νομοθετικές διαδικασίες μακροσκελέστερες και επομένως δεν έχουμε εμείς την ίδια δυνατότητα να κινούμεθα γρήγορα, τόσο γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος, όσο το Συμβουλίο. Γιατί πρέπει να τηρούμε τα προβλεπόμενα ημερολόγια των ολομελιών κτλ. Επομένως, η πρόταση αυτή μας επιτρέπει να μην αναλάβουμε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο και να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε πριν από το τέλος του μήνα. Είχαμε εξάλλου μία ανταλλαγή μεταξύ συντονιστών η οποία οδηγούσε στο συμπέρασμα μιας απλουστευμένης διαδικασίας. Αυτά μπορώ να σας πω ως πρόεδρος και ως εισηγητής. Ότι δηλαδή έχουμε την δυνατότητα μέχρι την 31η Οκτωβρίου να επανεξετάσουμε, αν θέλετε να το πούμε έτσι, τη θέση μας. Δηλαδή, χάρη ασφαλεία θα έπρεπε να πάμε σε απλουστευμένη διαδικασία. Αν όμω κατά αρκετά του υπόλοιπου μήνα δούμε ότι το Brexit δεν φαίνεται να λαμβάνει χώρα, θα μπορούσαμε, εγώ θα μπορούσα ως πρόεδρος της Επιτροπής, να αναβάλω την έκθεση για την πρόταση αυτή σε επόμενη ολομέλεια και επομένως εμείς ως Ρετζή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια εντελεχέστερη συζήτηση μεταξύ των συντονιστών και να προτείνουμε τροπολογίες για την ολομέλεια οι οποίες θα μας επέτρεπαν να τροποποιήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, τον κανονισμό. Επομένως, συμφώνως προς τα όσα αποφασίστηκαν από τους συντονιστές. και προκειμένου να είμαστε ασφαλείς σε περίπτωση που λάβει η χώρα η έξοδος σας προτείνω να υιοθετήσουμε σήμερα την απληστευμένη διαδικασία αλλά με τον αστερίσκο ότι θα μπορούμε να επανεξετάσουμε τη θέση αυτή και να μην διαβιβαστεί στην Ολομέλεια που είχε προβλεφθεί η πρόταση αλλά σε επόμενη ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούμε τις δικές μας προτάσεις τροπολογίας. Θα ήθελα λοιπόν τώρα πρώτα να δώσω το λόγο στους συντονιστές, μετά στα μέλη που θα ήθελαν το λόγο, γιατί πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που ε, καλούμαστε να λάβουμε εδώ σήμερα το απόγευμα. είμαι σίγουρος ότι μέσω της ανταλλαγής αυτής θα φτάσουμε στο σημείο είτε μέσω απλουσταμένης διαδικασίας είτε όχι να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Οι συντονιστές με τη σειρά παρακαλώ έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι υπέρ τη απλουστευμένη διαδικασία. Το είπα και στη συνεδρίαση των συντονιστών. Αλλά δεν θα πρέπει μόνο εξαιτία τη αμφιβολία αν θα αποχωρήσουν οι Βρετανοί, αλλά και εξαιτία το πώς θα κατανεμηθούν ε, ε, τα κονδύλια αυτά, 50% για τις ε, περιοχές που θα θυγούν από το Brexit. Η απόφαση στο Συμβούλιο είναι ξεκάθαρη. Το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να δώσει το 50% ε, από το Ταμείο Αλληλεγγύας ε, αλληλεγγύης και αυτό έχει κάνει και άλλες προτάσεις. Όσον αφορά την αποστευμένη διαδικασία, τότε θα πρέπει να δούμε και την πρόταση της Επιτροπής. Αν είχα παραπάνω χρόνο και εγώ θα προσπαθούσα να αντιρρυνήσω άλλες δυνατότητες ε, χρηματοδότησης, αλλά το 50% από το Ταμείο Αλληλεγγύης χωρίς ε, μεγάλες καταστροφές, το θεωρώ, στην που δεν πολύ μεγάλες καταστροφές, το θεωρώ παρόλα αυτά είναι αρκετά υψηλό ποσό. Και θα ήθελα να ξέρω αν θα μπορούμε τον των ε, να δούμε αν θα το εμποδίσει το Συμβούλιο και αν θα υπάρχουν άλλες προτάσεις για τη χρηματοδίτηση των περιοχών που θα πληγούν Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 5% που προβλέπετε θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλό. Merci, Andrei Novakov pour le groupe PPE. Novakov euh, για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Brexit είναι σαν τρενάκι του τρόμου. αν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να δώσει κάποια ελπίδα και να πει ψέματα για να φωτίσει το σκοτάδι που έχει πέσει πάνω από τον Brexit, α είναι έτσι. Όσον αφορά μας οι δικασίε που θα χρησιμοποιήσουμε, θα έλεγα ότι έχω επιφυλάξει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο, με μια απολυστευμένη διαδικασία κτλ. είναι ενδεχομένω θέμα άλλων διαδικασιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά θα πρέπει να ενεργήσουμε σίγουρα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε λιγότερο από ένα μήνα με ένα ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία. Επομένως, ανεξάρτητα τις ε, θέσεις που θα λάβουμε, άσχετα από τη διαδικασία, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πριν από την 1η ε, Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δηλώσει ότι στηρίζουμε αυτή την ταχεία διαδικασία με τα νέα δεδομένα για το Brexit, γιατί τότε το Brexit το, δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι μπορούμε, μπορέσαμε να, να δράσουμε με κάποια ταχύτητα, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος σίγουρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Λινάς. Ε, συμφωνήσαμε για την απλουστευμένη διαδικασία γιατί πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ε, και είμαστε στο ίδιο σημείο αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ε, ότι για τον Brexit οι ημερομηνίε δεν αλλάζουν. Αν κάτι αλλάξει, τότε θα αλλάξουμε κι εμείς. Αλλά μέχρι τότε είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε με ταχύτητα και με αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν τα χρήματα από το Ταμείο Λεγγύης νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα. Συμφωνώ λοιπόν, συμφωνούμε με την ε, γνώμη σα για την απροστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντονάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα Ιταλικά. Εγώ από την πρώτη στιγμή ήμουνα ο πρώτο συντονιστή που εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για την απλουσταμένη διαδικασία χωρί τροπολογίε. Για διάφορους λόγους. Καταρχάς για λόγους αρχής. Το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως θυμήσατε πρόεδρε, είχε προβλεφθεί για να καλύψει φυσικές καταστροφές και ατμοσφαιρικά φαινόμενα εν ώψη ή μάλλον συνεπία της έντονης κλιματικής αλλαγής που είναι όλο και πιο συχνά στις χώρες μας και επομένω επιφέρουν όλο και πιο σημαντικέ οικονομικέ ζημίε. Το να διατηρήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύη για τι φυσικέ καταστροφέ είναι υψηλωτά την προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανεί. Εξάλλου, οποιαδήποτε ζημία μπορεί να πορέει από no deal Brexit σχετίζονται με την ε, ελεύθερη αγορά και δεν έχουν καμία σχέση με φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Καθότι λοιπόν ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία η ελευθερία της αγοράς, η ελευθερία του ανταγωνισμού κτλ. είναι ύψιστα και κυρίαρχα δικαιώματα, το να επικαλούμεθα κάτι μάλλον το να χρησιμοποιούμε κάτι όπως τα διαδοτικά ταμεία αλληλεγγύης που είχαν προβλεφθεί για τελείως διαφορετικό σκοπό είναι στρέβλωση. Ως προς το επίγον του πράγματος είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν πάντοτε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μέτρων ευελιξίας για τις ε, συγκεκριμένες χώρες, ώστε και έναντι των προϋπολογισμών τους να εισαχθεί ένας χρυσός κανόνας ή οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο και να βρεθούν πόροι κονδύλια αλλού. Η προενταξιακή βοήθεια, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν πόροι του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως. Γιατί αν επιτρέψουμε απλουσταμένη διαδικασία αυτή τη στιγμή του να διάσουμε το 50% έως το 50% του ταμείου που είναι ταμείο αλληλεγγύης είναι επικίνδυνο προηγούμενο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον αντιστοίχω. Εγώ έχω αντίρρηση προς την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τοπολογίε. Επί τη ουσία θα μπορούσαμε Απλώ και μόνο να προτείνουμε να υποβάλουμε τροπολογίες για να περιορίσουμε το πόσο μπορεί να αδειάσει αυτό το ταμείο, όχι 50%, κάποιο μικρότερο ποσοστό ενδεχομένως, γιατί το 50% είναι οπωσδήποτε υπερβολικό και επί της ουσίας ε, μπορεί κανείς επ' αυτών, μάλλον με αυτές τις τροπολογίες υπόψη, να είναι υπέρ ή κατά κανείς. Επομένως, εγώ καθότι έχουμε τον κανόνα ότι πέντε μέλη μπορούν να μπλοκάρουν την όλη διαδικασία εφόσον δεν είναι υπέρ, καλώ τους συναδέλφους που συμφωνούν μαζί μου να εκφράσουν την διαφωνία τους ώστε να σταματήσουμε τη διαδικασία. ο συνάδελφος Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα είπαν διάφοροι συνάδελφοι σχετικά με τις περιπλοκότητες που υπάρχουν σχετικά με το Ταμείο αυτό. Προς μια κατεύθυνση επί της πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, αλλά ε, είναι εξαιρετικά συζητήσιμο το πόσο ευέλικτο θα μπορούσε να είναι το ταμείο, οι πόροι του ταμείου αυτού, αλλά αυτό που δεν μπορεί κανείς να συζητήσει είναι η απλουσταμένη διαδικασία, όπως είπε και η συνάδελφος. Πρέπει να καθορίζουμε με σαφήνεια ε, ποια είναι τα όρια, ποιε είναι οι κόκκινες γραμμές, ώστε να έχουμε εχέγγυα για αυτήν την όποια ευελιξία ή την όποια παραχώρηση. Επομένως, ήδη εγώ συμφωνώ επισήμως με την ε, κυρία Ντονάτο και θα είμαι μεταξύ των συναδέλφων που θα εκφράσουν την αντίρρησή τους για να μην επιτραπεί η αποσδεμένη διαδικασία Ευχαριστώ. Την... Ε, τώρα το λόγο έχει από την Ευρωπαϊκή Αν κατάλαβα καλά, τον πρόεδρο προτείνει αυτή τη στιγμή ε, μία διπλή διαβάθμιση για να είμαστε ευέλικτοι στη διαδικασία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα πώς θα, ε, ποια θα είναι η έκβαση του Brexit, αν θα υπάρξουν συμβασμοί Και, τα λοιπά. και γι' αυτό το λόγο, όπως και η συνάδελφος από τους Πράσινους, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την αντίδραση σε δύο διαφορετικά επίπεδα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφορετική τροπή και να χρησιμοποιήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία και να δούμε αν θα έχουμε τελικά χρόνο, στην οποία περίπτωση θα μπορέσουμε ενδεχομένως να επιστρέψουμε στις άλλες διαδικασίες και γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση του Προέδρου. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Ε, ζητούν το λόγο η κυρία Κρέτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Θα μιλήσω στη μητρική μου. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να προσθέσουμε τα κράτη-μέλη Ξέρουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι ο μεγαλύτερος πληρωτή στην Ευρωπαϊκή, στον Ευρωπαϊκό ε, Προπολογισμό με 13% και η πολιτική συνοχής είναι το 75% του προπολογισμού. Θα ήταν πολύ ε, κακό για συγκεκριμένε περιφέρειες και κράτη-μέλη αν ε, έχουμε ένα Brexit ατακτό Υπάρχουν πολλές, ε, πολλά έξω που πρέπει να καλυφθούν το 2020 σε αυτές τις ε, περιφέρειες και αν τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρέωση να συμμετέχει στον προπολογισμό στο 2023. Υπάρχει το ρίσκο να μην πάνε τα χρήματα αυτά στις ε, περιφέρειες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Κατά δεύτερον, όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, συμφωνώ με την συντονίστριά μας και με σας κύριε Πρόεδρε. Το Ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο που δημιουργήθηκε για έκτακτες περιστάσεις. Τα τελευταία τελευταία χρόνια είχαμε πολλά προβλήματα με φυσικές καταστροφές όπως τον σεισμό στην Ιταλία και υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν τις αποδείξεις τις σχετικές για τις φυσικές καταστροφές και στο τέλος ε, πολλές φορές συμβαίνει να μην είναι παρακεί τα κονδύλια αυτά. Οι πυρκαγιές στην Πορτογαλία χάθηκαν πάρα πολλές ζωές. Στο τέλος όμως αυτό που υπόθηκε ήταν ότι, ότι ε, ήταν μόνο ε, οικονομικές καταστροφές και δεν, παρα, ε, δεν παρασχέθησαν άλλες αποζημιώσεις. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν το ταμείο αυτό, κυρίως για τις φυσικές καταστροφές. Ευχαριστούμε την κυρία Κρέτο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπόκοβιτς. Εφόσον μιλάμε για το Brexit και για τις φυσικές καταστροφές, στις φυσικές καταστροφές και στην κλιματική αλλαγή πιστεύουν ε, κάποιοι ακόμα ότι δεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά για τον Brexit αυτό είναι ξεκάθαρο φυσικά. Εγώ υποστηρίζω την αλληλεγγύη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλληλεγγύη με αυτούς που ε, έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα. Φυσικά το Brexit θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς. Το ποσό που προβλέπετε εδώ είναι πολύ χαμηλό. Ο Τζόνσον κάνει λόγο για 80 δισεκατομμύρια. Από την βρετανική πλευρά μιλάμε για 600 εκατομμύρια μέσα σε 1,5 χρόνο και το αποθεματικό που υπάρχει θα πρέπει ε, αφορά κυρίως ε, ε, τις φυσικές καταστροφές και ναι, με θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό, αλλά θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να ενεργήσει πολύ γρήγορα, ακόμα και θα πρέπει αργότερα να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες για να καθισχάσω αυτούς που φοβούνται ε, ότι θα υποστούν πολύ μεγάλες βλάβες από το Brexit σε αυτά τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν οι σκέψεις των 0,3% του ΑΕΠ ε, θα μειωθεί και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια, μια διαφορετική διαδικασία είναι καλό, επομένω να δώσουμε ένα σήμα ε, ως προς όλα αυτά για αυτούς που ε, ε υποστηρίζουν το πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ριμπό. Κύριε Πρόεδρε, Όσον αφορά αυτή την απλουστευμένη διαδικασία, θα πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα σε μια κατάσταση που θα συμβεί και που θα είναι καταστροφική για πολλές χώρες. Και η χώρα μου ανήκει σε αυτές. Έχουμε και προηγουμένω συζήτησαμε για το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Τώρα όμως έχω πέντε λεπτά εκ μέρου ε, του κράτους μου και άλλων κρατών στο Συμβούλιο να μεταφέρω την παράκληση να ελέγξουμε το θέμα αυτό, να δούμε ποια κράτη-μέλη θα δεχτούν περισσότερο από το Brexit. Και αυτά είναι η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία. Και ότι αυτά τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτά τα ταμεία, από τις αυτού του ταμείου. Θα ήθελα λοιπόν να το ελέγξουμε ξανά το κείμενο, να προτείνουμε τροπολογίε γιατί βρισκόμαστε στην κατάσταση που πλησιάζει η 25 Οκτωβρίου και η λύση είναι η απλουστευμένη διαδικασία, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένω να κάνουμε και κάτι άλλο πιο επικοδομητικό, η απλουστευμένη διαδικασία, αλλά και η απλουστευμένη διαδικασία με τροπολογίες είναι ένα ενδεχόμενο ως το τέλο του μήνα. Είναι και, αυτή, είναι αυτό ένα ενδεχόμενο. Γιατί αν κάποιο είναι ενάντια σε αυτή την προσέξη μπορεί να προτείνει τροπολογίε. αλλά θα έχουμε ένα κέρδο χρονικό. Ο Μπόρι Τζόνσον δήλωσε, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι ό,τι και να γίνει, ο κόσμος θα χαλάσει, αποχωρούμε στο τέλο του μήνα. είναι στενό το χρονικό πλαίσιο, να το τηρήσουμε, αλλά παράλληλα να έχουμε και αυτή την ευελιξία για να εκφράσουμε την άποψή μας και επομένως να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία ως μια συμβαστική λύση μεταξύ όλων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, λίγο Έχω ακόμα δύο μέλη στον κατάλογο των ομιλητών και θα κλείσω μετά. Κοτζολίνο και μετά ε, ο φίλος του Φίντε. Ε, πρόεδρε, η τελευταία πρόταση που έγινε μου φαίνεται πιστική. Να έχουμε δηλαδή απλουστευμένη διαδικασία, αλλά με τροπολογίε εδώ στην Επιτροπή, δηλαδή να έχουμε το χρόνο προπαρασκευή εν ώψη τη Ολομέλεια. Και επειδή, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είπαν ότι δεν είμαστε ομόφωνοι εδώ. Δηλαδή, την ώρα που εμεί θα πάμε σε απλουστευμένη, το Συμβούλιο θα μπορούσε να πάει σε διαφορετική κατεύθυνση και να υποσκάψει την προσπάθειά μα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πρόταση ώστε να συμφωνούν όσο το δυνατόν οι περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά και εγώ θα συμφωνούσα ότι υπάρχουν άλλες γραμμές του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κονδύλια για τέτοιου είδους περιπλοκές. Και όχι αναγκαστικά αυτό το ταμείο ανάλογα με το τι θα συμβεί και στο τέλο του μήνα. Ευχαριστώ. Λέει Πάνσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι απολύτω απαράδεκτη αυτή η διαδικασία πρόταση χρησιμοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Λεγγύης που το χρησιμοποιούμε ως ATM επειδή απλώς δεν λάβαμε τις αποφάσεις που έπρεπε να λάβουμε. Τις προβλέψεις δηλαδή που έπρεπε να γίνουν εν ώψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που μπορεί να λάβει η χώρα στο τέλος του μήνα που είναι αύριο το απόγευμα, σε να λέμε. Ε, δηλαδή ο αντίκτυπος του προβλήματος αυτού ήταν σαφής. Θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη. Το να χρησιμοποιούμε το ταμείο αυτό σαν να είναι ATM και βάζουμε την κάρτα και τραβάμε χρήματα, θα ήταν ένας τρόπος, μια επιλογή εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι αποθεματικό, γιατί αν συμβεί απόψε, αύριο, μια πλημμύρα, ένα σεισμός, χτυπάω ξύλο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Κανείς δεν διαφωνεί ότι το Brexit θα δημιουργήσει προβλήματα, δύσκολα προβλήματα και δυσκόλως μετρήσιμα έναντι τι να σας πω τώρα για να πω το τυχαίο παράδειγμα γέφυρας που ξαφνικά καταραίει και τότε μπορείς να κάνεις εκτίμηση της ζημιάς. Και υπό την έννοια αυτή, όπως είπε και ο κύριος Κοτσολίνο, ε, πρέπει να έχουμε μια ακριβέστερη εκτίμηση πρόταση. Εμείς πρέπει λοιπόν να αρνηθούμε την απλουστευμένη διαδικασία γιατί υπάρχει αλανθασμένη αρχική επιλογή κατεύθυνση χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών. Σα ευχαριστώ, λέει ο Ε, να πω και εγώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ ότι δεδομένη της κλιματική αλλαγή των καιρικών φαινομένων, των φυσικών καταστροφών που είναι πιθανόν να λάβουν χώρα, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε δυνατότητα να δρούμε, να αντιδρούμε ταχαίως και πλήρως. Επί τη βάση των απόψεων που ακούστηκαν εδώ, το 52-2 του ιστορικού κανονισμού είναι πολύ αμφίβολο να οδηγήσει σε λύσεις μέσω της απλουστομένης αυτής της διαδικασίας και της ακόλουθης υποβολής τροπολογίων θα πρέπει εμείς ε, δηλαδή, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε, με ευέλικτο τρόπο ανάλογα με το τι μπορεί να μας προκύψει και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι ο προτινόμενος τρόπος. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση της σημερινή. Δεν αναφέρομαι στην ειδική μου υπηκότητα πάρα πολύ συχνά, αλλά εκπροσωπώντας την Νότια Ιρλανδία, Νομίζω ότι πράγματι είναι η κατάλληλη στιγμή να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τους βόρειους γείτονές μας και αναγνωρίζοντας τις περιπλοκές της αποχώρησης που είναι πρώτων πυλών. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τους συμπολίτε μας που ζουν πάρα πολύ κοντά σε μας στο Διβλίνο δεν είναι φυσική καταστροφή, συμφωνώ, είναι ανθρώπινη τεχνητή καταστροφή, αλλά την ανθρώπινη χείρα τη βλέπουμε και στις φυσικές καταστροφές μέσω της κλιματικής αλλαγής και μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Επομένως, υπό μια κάποια έννοια θα μπορούσαμε να το προεκτείνουμε και στην κάλυψη της τεχνητής αυτής καταστροφής. Ευχαριστώ. Ε, η συνάδελφος είχε ζητήσει το λόγο και κλείνω μετά τον κατάλογο όμω. Ε, dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να επιδείξουμε εδώ αλληλεγγύη και θα πρέπει να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις χώρες εκείνες που θα είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο τον οικονομικό και τον λοιπό αντίκτυπο έναντι της, ε, άτακτης, ε, της πιθανότητας άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασίλειου τώρα ως προς το ταμείο το συγκεκριμένο ταμείο και το κατά πόσον μπορεί να θεωρηθεί ως ε, μέσο βάση θεμέλιο όπως σωστά είπαν οι συνάδελφοι αυτό το ταμείο είχε προβλεφθεί για να αντιμετωπίσει διάφορα φυσικά φαινόμενα καιρικά φαινόμενα ε, ακραίες καταστροφές, έκτακτες ανάγκες δηλαδή αυτού του είδους. Τώρα εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος άλλου είδους ακραίων φαινομένων και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Πιστεύω ότι μπορούμε εδώ να προβλέψουμε απλουσταμένη διαδικασία με, δυνατότητα, τη δυνατότητα υποβολής τροπολογιών. Je pense que la, la responsabilité euh, politique oblige euh, Υποχρονόμαστε να, ε, ε, να προβλέψουμε. Για ακόμα και αν ε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την υπόθεση, ίσως υπάρξει ένα σκληρό Brexit την 31η Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να, να αντιμετωπίσουμε και αυτή την προοπτική. Ο διάλογος όμως, ε, η συζήτηση ε, δείχνει ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός όσον αφορά στην ε, πρόταση έτσι όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια απροθυμία για την απλουστευμένη διαδικασία και και εγώ θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, είμαι μεταξύ αυτών που θεωρεί ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεισφέρει και να, α, ως συνομοθέτης να πράξει το ρόλο του. Δεν, δεν θέλω να βρίσκεται η Επιτροπή σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε όμως την υποχρέωση επίσης ε, να ε, φανταστούμε αυτό που ε, είναι ίσως πιθανότητα 31 Οκτωβρίου, ένα σκληρό Brexit. Η απροθυμία ε, ε, σχετίζεται με τον πυρήνα της πρότασης. Το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, είναι ένα ταμείο που προορίζεται για την αντιμετώπιση κλιματικών, φυσικών καταστροφών και η πρόταση που παρουσιάστηκε χρειάζεται τουλάχιστον κάποιες ε, τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας προτείνω χωρίς να μπούμε σε διχαστικές ψήφους, να βρούμε μία λύση συμβιβαστική. Η συμβιβαστική λύση, όπως ε, μας υπενθύμισε ο κύριος Μπιζού, μία από τις συμβιβαστικές υπάρχει στον κανονισμό. Ο κανονισμός λοιπόν προτείνει ότι ο πρόεδρος σε μια απλουστευμένη διαδικασία, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει ο ίδιος ή ο εισηγητής να συντάξει μια σειρά τροπολογιών βάσει της συζήτησης της Επιτροπής. Εάν υπάρξει ε, ελάχιστος αριθμός ε, τότε εγκρίνεται η ε, τοπολογία και παρουσιάζεται στην Επιτροπή. Αυτό είναι μία πιθανότητα, δηλαδή έχουμε μία επλουστευμένη διαδικασία μαζί με, τροπο, τροπολογίες. Το κάναμε στην Επιτροπή αυτή για όσους από εσάς ήσασταν την προηγούμενη νομοθετική περίοδο και αυτές μάλιστα ήταν πραγματικές ε, τροπολογίες ε, που προέρχονταν από την ε, ολότητα της Επιτροπής μας. Υπάρχει μια άλλη, ένα άλλο υποθετικό σενάριο, ότι έστω ότι εγκρίνεται σήμερα η απλουστευμένη διαδικασία, όπως σας προτάθηκε, όπως περιουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, όπως βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση, τότε ζητάμε ε, την, ε, να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια και ω ε, ως τότε θα εξετάσουμε τις τροπολογίες που θα εξεταστούν στην Ολομέλεια κατά την ψήφιση του κανονισμού. Ίσως η πρώτη λύση είναι μία που, ε, με την οποία συμφωνούν όλε οι πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να ε, ανοίξω εκ νέου την ε, συνάντηση για τους συντονιστές. Αν θέλετε λίγο χρόνο, μία μικρή παύση πέντε λεπτών, τότε σας την παραχωρώ. Αλλιώς ξεκινάει η συζήτηση και δίνω το λόγο στους συντονιστές οι οποίοι εξέφρασαν ε, την ε, αντίρρησή τους γιατί δεν θα έπρεπε να εγκριθεί η πρόταση. Τον λόγο έχει ο κύριος Νοβάκοφ. Θα ήθελα ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Πολύ καλά. Έχετε πέντε λεπτά. Επανερχόμαστε σε πέντε λεπτά Έχουμε πέντε λεπτά καιρό Τα πέντε λεπτά αυτά ελπίζω να ήταν χρήσιμα και παραγωγικά. Τώρα επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τους συντονιστές. Θα ήθελα να τους ζητήσω να μας παρουσιάσουν με σαφήνεια τις προτάσεις τους ε, και μετά θα θέσω σε ψηφοφορία μία πρόταση ζητώντας εάν λοιπόν ε, είναι η απλουστευμένη, ψηφοφο... Ε, απλουστευμένη διαδικασία, αν... θα ζητήσω αν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Ο κύριος Νοβάκοφ από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η θέση του κόμματο, της ομάδας μας ε, είναι η ίδια. Ε, υποστηρίζουμε την, το 52,2, όμως υπάρχουν πέντε μέλη που αντιτίθενται. Αλλά ε, η πρόταση είναι να, να κρατήσουμε το 52,2. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας ε, θα είναι έτοιμη να ακολουθήσει την ε, πλουστευμένη διαδικασία. Δηλαδή και εμείς συμφωνούμε με το 52,2. Ο συνάδελφός μας, ε, κύριος Κνοτέκ, και εμείς υποστηρίζουμε την πλουστευμένη διαδικασία με, την, με τις πιθανές τροπολογίες. Δηλαδή Είμαστε υπέρ του 52,2. Ευχαριστούμε πολύ ε, για τους πράσινους. Ε, συμφωνούμε με την πληστοποιημένη διαδικασία με τις τροπολογίες, αλλά θέλουμε να ε, μάθουμε πώς θα φτάσουμε στις τροπολογίες, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα απλά να, να προταθούν τροπολογίες, θα πρέπει να εκπροσωπήσετε την Επιτροπή. Ευχαριστώ από την ομάδα ΙΔΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, αντιτιθέμεθα στην, με την διαδικασία προστευμένης, ε, την προστευμένη διαδικασία, γιατί ακόμα και σε αυτή την ε, περίπτωση δεν έχουμε την δυνατότητα ε, να καταγράψουμε τις ε, τροπολογίες και να τα συζητήσουμε όπως ε, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς. Την απορρίπτουμε λοιπόν. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα φέρει καινούργια πρόταση με ένα άλλο ταμείο και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από το, η ομάδα των μεταρρυθμιστών είναι υπέρ το, του συμβιβαστικής λύσης. Επομένως, ε, είμαστε υπέρ μιας απλουστευμένης διαδικασίας με τροπολογίες. Όχι, Πρόεδρε, διότι είναι προφανές ότι υπάρχει μία αντίφαση. Ακούσαμε από διάφορους συναδέλφους επικρίσεις για τις επιλογές της Επιτροπής, της Επιτροπής με του Ταμείου αυτού, ε, μέσω τροπολογιών θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε, να δείξουμε προς άλλο ταμείο. Είπαμε πριν, αλλά ακούμε ιδιαίτερα αντιφατικά σημεία σε σχέση με αυτά που άκουσαμε αμέσως πριν και τη διαδικασία που φαίνεται τελικά να υποστηρίζει. Γιατί αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε απλουστευμένη διαδικασία με τις τροπολογίες έτσι όπως τις προτείνατε Πρόεδρε και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς ε, η, τελικός, η τελική θάση θα είναι επί της ουσίας και όχι επί της πλειοψηφίας θα πρέπει μέσω τροπολογιών να εκφράσουμε τις θέσει μας. Το απλούστερο θα ήταν να καλέσουμε την Επιτροπή να επανυποβάλει διαφορετική λύση με μέσα που θα είναι καταλληλότερα για το θέμα αυτό. Ώστε να μπορούμε να έχουμε απλουστεμένη διαδικασία τότε πλέον χωρίς κανένα πρόβλημα. Η θέση μας δεν έχει διαφοροποιηθεί, επομένως, Πρόεδρε, λυπούμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για την ε, αριστερά. Μη υπέρ τη απλουστευμένη διαδικασία με τροπολογίε. Προσβλέποντα ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να εκφράσουν την άποψη της, πλειοψηφ πια. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Στο ECR να πω ότι ε, αντιλαμβάνομαι απολύτως την τοποθέτησή σας. Όμως πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εάν η απλουστευμένη διαδικασία με τροπολογίες δεν εγκριθεί, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν θα εξεταστεί η πρόταση. Γιατί τότε θα έχουμε τακτική διαδικασία επί τη βάση της πρότασης όπως υπευλήθη από την Κομισιόν. Από εκεί πέρα υπάρχουν τροπολογίες που θα μπορούσαν να υποβληθούν για την απόρριψη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά θα πρέπει όμως και εδώ και στην Ολομέλεια να υπάρξει πλειοψηφία. Εγώ είπα ευθύς εξ αρχής ότι κανείς στην Επιτροπή μας δεν είναι κατενθουσιασμένος με την πρόταση αυτή. Πρόταση που έχει διάφορα κενά και διάφορες ελλείψεις. Η οποία όμως δείχνει να ανταποκρίνεται σε μια δυνητική επίγουσα ανάγκη. Επομένως, έχουμε και εμείς την ευθύνη να λειτουργήσουμε σε μια υπόθεση εργασίας ε, ενός no deal και να δούμε σε αυτό το πλαίσιο ποιος θα είναι ο ρόλος μας και υπ' αυτές τις προϋποθέσεις να υποβάλουμε τροπολογίες. Λοιπόν, έχοντα ακούσει τις ομάδες, έχουμε εδώ μια πρόταση, Απλουστευμένη διαδικασία. λοιπόν, επί τη βάση του άρθρου 52, παράγραφος 2 του κανονισμού, με τροπολογίες της Επιτροπής οι οποίε βεβαίω θα αποτυπώνουν τις διάφορες πολιτικές ομάδες, τις θέσεις τους, και που θα τις επεξεργαστεί το προσωπικό των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει αντίρρηση έναντι αυτής της πρότασης έτσι όπως την είπα. Αν έχουμε αντίρρηση παρακαλώ εκφραστείτε. Αν θέλετε απλώς σηκωθείτε όσοι έχουν αντίρρηση. Μάλιστα. Έξι μέλη λέει ο πρόεδρος, επτά είναι τα μέλη που έχουν αντίρρηση, τα πέντε επαρκούν και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διαδικασία τακτική. Και επομένως αύριο θα επανεξετάσουμε το θέμα στους συντονιστές. Άρα μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, το οποίο αφορά στον κατεξιοδότη συγκανονισμό που συμπληρώνει, με που συμπληρώνει τον κανονισμό για την καταποκοπή χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ένα σύστημα χρηματοδότησης και τεχνικής αρρωγής για τα έργα κατεξιοδότηση υπό το άρθρο 67 παράγραφος 5b του κανονισμού κοινή διάταξη που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να προβλέπει κατά χρηματοδότηση. Και τότε ο κατεξιδότης είναι κανονισμός προβλέπει τέτοιο κατά ποσό για την τεχνική βοήθεια που θα μπορεί να δοθεί στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή λέει ότι η τεχνική αυτή αρρωγή ε, βοηθείται ιδιαίτερα από την απλούστευση δεδομένων των θεματικών, των αντικειμένων δηλαδή της τεχνικής αυτής βοήθειας και του αριθμού των δικαιούχων. Λοιπόν, τα ποσά που προτείνει η Κομισιόν είναι για το ΦΕΝΤΕΡ εκτός εδαφικής συνεργασίας FSE, FC, FEADER 4% για το FEAM και FEDER εδώ έχουμε εδαφική συνεργασία 6% η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων που θα υποβληθεί ως ψήφος στην Ολομέλεια προβλέπεται για τις 28 Οκτωβρίου του 2019. Και θα καλούσα τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει το σχέδιο κατεξιοδότηση κανονισμού της και θα δώσω ακολούθως το λόγο στα μέλη. Παρακαλώ την στους προσώπους της Κομισιόν. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μας παρουσιάσατε την πρόταση. Πολύ ολοκληρωμένα παρουσιάστηκε η πρόταση. Λίγα θέματα θέλω να θίξω. Ο κανονισμός που μας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγουμε, ε, να χρησιμοποιήσουμε τις καταποκοπή πληρωμές και περισσότερη απλούστευση γενικά στην εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής. και ως μέλος ε, της Επιτροπής για την περίοδο 2020-2023 έχουμε εισαγάγει ήδη απλουστεύσεις όπως και την ε, καταποκοπή χρηματοδότηση για την τεχνική υποστήριξη. Αυτό παρέχει λοιπόν και μία γέφυρα ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και την προγραμματισμένη προσέγγιση για την επόμενη περίοδο. Δίνει τα για προγράμματα να χρησιμοποιήσουν την καταποκοπή πληρωμή για τεχνική στήριξη τεχνική υποστήριξη είναι μια από τις βασικές, ένας ε, από βασικούς τομείς για τέτοιου υποστήριξη, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοια προγράμματα και έχουν ως σκοπό ε, την διευκόλυνση των προγραμμάτων, της εφαρμογής τους ε, και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η τεχνική στήριξη γίνεται η οργάνωση για τους δικαιούχους, για τους οργανισμούς, για τις προκηρύξεις, τις ε, συνεδριάσεις, την εφαρμογή των προγραμμάτων και γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή της τεχνικής στήριξης ε, περιέχει και μεγάλο διοικητικό άχθος ε, στις αρχές και στους δικαιούχους και αυτό περιλαμβάνει πολλές φορές ελέγχους από εισιτηρία, από μικρές δαπάνες, όλα από τα οποία αποτελούν ε, τακτικά, τακτικές πρακτικές σε τέτοιες διαδικασίες. Προτείνουμε λοιπόν μια πολύ απλή επιλογή την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα και συνδέουμε την ε, παροχή τεχνικής υποστήριξης μαζί με την εκτέλεση και την πρόοδο. Επομένως, όταν υπάρχουν αιτήματα για πληρωμές, εντοπίζουμε τα ποσοστά που ορίζει ο Πρόεδρος για κάθε ε, τομέα και συμπληρώνουμε με το αντίστοιχο ποσό στην πορεία του έργου. Δεν σημαίνει ότι αυτό χρειάζεται περισσότερο περισσότερα κονδύλια, γιατί αυτά καθορίζονται στον κανονισμό κοινών διατάξεων. Και φυσικά η τεχνική στήριξη είναι συγκεκριμένη. Αυτό όμως που αφαιρείται είναι το διοικητικό άχθος στη διαχείριση της τεχνικής στήριξης, των ελέγχων επαλήθευσης και επιτρέπει παράλληλα τις ε, αρχές τις διευκολύνει να παρέχουν υψηλής ποιότητας ε, προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ για την σαφή παρουσίαση. Τον λόγο έχουν οι συντονιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, για την πρόταση καταξιδοτότηση πράξης. Χρειάστηκε και πολύ συζήτηση. Ήμουν εισηγήτρια εγώ για το Omnibus. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία από την πλευρά της Επιτροπή μας να γίνει αυτή η αλλαγή ε, στην απλούστευση και την κατάρριξη της ε, γραφειοκρατίας στην πολιτική συνοχής. Είχαμε εντατικές διαπραγματεύσεις και το σημαντικό για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες είναι αυτή η απλούστευση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τρέχουσα περίοδο. Επομένω, είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση καταξιοδότηση πράκτη από την Επιτροπή, ώστε οι διαδικασίε να μπορέσουν να προχωρήσουν χωρί μεγάλε δυσκολίε και χωρίς αλλαγή επιχειρησιακών προγραμμάτων ή εταιρικών σχέσεων. Και φυσικά για αυτό το λόγο υποστηρίζω αυτή την πρόταση και προτείνω το στομότερο δυνατόν να την θέσουμε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νοβάκοφ Έχω ένα ιστορικό για την καταπολέμηση ε, γραφειοκρατίας. Ε, θα ε, υποστηρίξω λοιπόν την διευκόλυνση της ζωής των δικαιούχων. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση. Είναι μια πρόταση που κοιτάει μπροστά, ειδικότερα σε σχέση με, την, με τον επερχόμενο κανονισμό, κανονισμό κοινών διατάξεων. Ο στόχος είναι η απλούστευση θεωρώ ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να δίνουν λιγότερο διοικητικό φορτίο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να αποδεχθεί, να εγκρίνει την πρόταση του, ε, του, του Κοινοβουλίου για την διανομή κονδυλίων για τεχνική ε, βοήθεια. Λοιπόν, θα πρέπει να αυξηθεί κατά το ποσοστό των κονδυλίων που διτεύεται για τεχνική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν το λόγο τώρα το, η ομάδα Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δικαιούχοι ζητούν την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού άχθους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή για, την κατεξουσιοδότηση, για τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η πράσινη Ευχαριστούμε. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή. Προσμένουμε σε αυτή την κατεξουδότηση πράξη. Ε, συνεχίζουμε τώρα με την ομάδα ΙΔΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρ αυτής της κατεξουδότησης πράξης γιατί αυτή η απλούστευση είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο ώστε να μπορέσουμε να αναμειώσουμε το διοικητικό άθος και να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τους δικαιούχους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να την επικροτήσουμε ε, ως πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ οι συντονιστές του, της ΓΟΕ και του ΣΕΣΑΡ δεν είναι παρόντες, δεν υπάρχουν ειδικέ αντιρρήσεις, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, ότι η εξέταση λύγει εδώ. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι και θα ήθελα να απευθυνθώ μάλιστα και στην Επιτροπή ότι η συζήτηση που είχαμε για το ζήτημα της ε, πλουστευμένης διαδικασίας, αν θα την υιοθετήσουμε ή όχι λοιπόν, ε, στην πραγματικότητα όλα όσα υπόθηκαν από το σύνολο δείχνουν εδώ ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ρέτζη ε, δεν θέλουν να ασκήσουν βία. Θέλουν την βελτίωση των πραγμάτων, πρέπει ε, λοιπόν ε, ως συνομοθέτες ε, να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο μας στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Μένουμε προς το παρόν εδώ. Σε λίγο, στις 6.30 θα ξανασυναντηθούμε για την ακρόαση της ε, Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Θα δώσουμε ραντεβού στην ε, αίθουσα Γιάν 2Q2 Σας ανακοινώνω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις 4 Νοεμβρίου από τις 3 η ώρα μέχρι τις 6.30 και 5 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν. Merci. Ευχαριστούμε τους Διερμηνείς για την συνεισφορά της για την συνεισφορά τους στην ε, ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε πολύ.